Και συνεχίζουμε στην ημερήσια διάταξη με την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις μελλοντικέ νομοθετικές προτάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ε, πρόκειται για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Από εκεί προέρχεται η ερώτηση αυτή. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Sharon που είναι ε, εκείνη που έχει συντάξει την ερώτηση αυτή. Ο Επίτροπος Ρεν θα απαντήσει στην συνέχεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Μπόλιτς, παρακαλώ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Επίτροπε. Πρόκειται για την απάντηση της Επιτροπής ΕΚΟΝ στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα και τους μηχανισμούς σύγκλησης. Πρώτα απ' όλα έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο για τη μακροοικονομική διακυβέρνηση με τη δέσμη 2 και 6 οδηγιών. Επίσης ως προς την Τραπεζική Ένωση αρχίσαμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα με το, τη δέσμη 6 οδηγιών, το six ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σημειώσει πρόοδο και εμείς σας πιέζουμε και η αντιπροσωπεία της ΕΚΟΝ άκουσε τα, ίδια σχόλια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, πέρσι. Πρέπει να υπάρξει όμως ε, κατανόηση σε σχέση με αυτά που ήδη έχουμε κάνει για να ε, τύχουμε δίκαιη μεταχείριση. Βεβαίως έχει έρθει η στιγμή να εφαρμοστεί σωστά ε, το, η δέσμη των 8 οδηγιών, το 6 pack και το ΤΟΥΠΑΚ, δηλαδή ταυτόχρονα με νέες ιδέες. Χρειάζεται σαφήνεια σε σχέση με την προστιθέμενη αξία που θα προσέφερε αυτό σε σχέση με την κειμένη νομοθεσία. Μήπως θα έπρεπε τους τελευταίους 18 ε, ε, να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί και να μην υπερβάλλουμε και να αρχίσουμε να μιλάμε ήδη για τη δέσμη των 10 οδηγιών. Ε, πάντως, σε, από όλους τους παρατηρητές σχολιάζεται το ότι χρειάζεται η Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι σε μια αλληλέγγυα οικονομία όπου υπάρχει λογοδοσία. Όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις σημειώθηκε έλλειψη διαφάνειας, διακυβερνητισμός ε, ανάμεσα ε, στα διάφορα κράτη-μέλη και διενέξεις ε, ανάμεσα τους. Γνωρίζω ότι επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κοινοτική μέθοδο και όχι τον τη διακυβερνητική προσέγγιση. Θα σας υποστηρίξουμε, όμως έχουμε ήδη μια πανοπλία διοικητικών μέτρων και έχουμε απομακρυνθεί από τους πολίτες. Ας μην επιδεινώσουμε την κατάσταση. Έχουμε την τον εξάντε συντονισμό επίσης. Η πρώτα πρότασή σα δεν διευκρίνησε την προστιθέμενη αξία ε, τη ε, προτινόμενη δρυξικέλευτη πρόταση ε, στο βαθμό που έχουμε την Ευρώπη 2020, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το Ταμείο συνοχή τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το κάθε εξή. Και για να επιδεινωθεί η κατάσταση, η Επιτροπή ΕΚΟΝ ζήτησε ρητά η αδίποτε νέα διάταξη να ενταχθεί στι διατάξει περί Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να έχουμε απόλυτη διαφάνεια και κοινοβουλευτικό έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μεταβατικές διατάξεις ε, για τη μεταφορά νομοθεσίας από το ευρωπαϊκό προς το εθνικό επίπεδο, ούτω ώστε να είναι ομοιόμορφη η εφαρμογή. Εμείς προτείνουμε κώδικα σύγκλησης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση μεταγράφεται σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας ε, για να έχουμε συγκεκριμένα κίνητρα ω προς τις συμβατικές υποχρεώσεις ε, οι οποίες όμως ε, ε, δεν πρέπει να προβλεφθούν για τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Μια συνεργατική διαδικασία χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά προβλήματα. Τα ταμεία και τα κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν θα μπορούν να αποτελέσουν έναν εμβριακό κοινοτικό προϋπολογισμό που θα αντιμετωπίζει τα ασύμετρα σοκ στην οικονομία. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε περιεχόμενο του πακέτου. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική δέσμευση για ε, περαιτέρω εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε στον τύπο όλων των χωρών ότι όλοι επιζητούν την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τα ταμεία CCI εκτό όμω του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού, εκφεύγοντας έτσι οδήποτε κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και πέραν αυτού, ε, χρειαζόμαστε λεπτομερέστερε προτάσει σε σχέση με το πώ ένα νέο όργανο σε σχέση με το αν θα πρέπει να υπάρξει και υπό ποια μορφή θα πρέπει να υπάρξει. Αν λοιπόν θα καλυφθούν όλε οι χώρε, είτε είναι στην ε, Ευρωζώνη είτε όχι, είτε ε, ε, υπάρχει μνημόνιο είτε όχι, να δούμε ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία. Ο εξάντε συντονισμό και η λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίση θα πρέπει να εδράζονται επικρατεών στατιστικών στοιχείων σε σχέση με τον δημοσιονομικό συντονισμό συντονισμό των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε ενοποιημένα στατιστικά στοιχεία για του ετήσιου λογαριασμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών μελών καθώ και των ΟΤΑ, των αρχών τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, θα πρέπει να περάσουμε ε, αυτό το ηχηρό μήνυμα εάν δεν κατοχυρώσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο από το Κοινοβούλιο που είναι συνομοθέτη και συναρχή εκτέλεση του προπολογισμού. Δεν μπορούμε να δεχθούμε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση. Σα ευχαριστούμε κυρία Μπόλ. Τώρα θα ακούσουμε τον Επίτροπο Ρένα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει την κυρία Μπόλ. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, καλή σας ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροφή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ερώτηση όσον αφορά τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ. Πρόκειται για διορθωτικές μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Προφανώς και χρειάζονται τέτοια νέα μέτρα. Έχουμε ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αναφίβολα χρειάζεται περισσότερη δουλειά, όπως ακριβώς υπογράμμισε και η κυρία Μπόλς. Πρώτα απ' όλα, ο οικονομικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί. Η Τραπεζική Ένωση θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που είναι πολύ βασικό για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Άλλα σημαντικά στοιχεία για την βελτίωση της οικονομικής ολοκλήρωσης αναφέρονται στις δύο ανακοινώσεις που παρουσιάσαμε τον Μάρτιο. Πρόκειται για τον συντονισμό των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και για τα μέσα συντονισμού και ανταγωνιστικότητας. Επιτρέψτε μου εδώ να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στη φύση των ανακοινώσεων αυτών. Πρόκειται για ιδέες όσον αφορά τα συστήματα που ισχύουν. Βάση και προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των χωρών μελών, των διάφορων εμπλεκόμενων, και Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις αυτές τις εξετάζει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο συγκεκριμένα θα ενημερωθεί πλήρως για την διαμόρφωση πρωτοβουλειών που θέλουμε να πάρουμε σύμφωνα με τις συνθήκες. Πέραν αυτού, για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο και να καλύψει και τις πρωτοβουλίες αυτές. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή θα συζητήσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν ώψη των συμπερισμάτων του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης μπορεί να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων για τις σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις ώστε να εξηγήσουν τις θέσεις τους. Έτσι θα υπάρξει έλεγχος. Για την ερώτησή σας τώρα όσον αφορά την σχέση των ε, ανακοινώσεων αυτών με τον συντονισμό και την διακυβέρνηση, πρέπει να ξέρετε ότι ο εξόντε συντονισμός έχει να κάνει με τις μεταρρύθμισεις και βασίζεται στο άρθρο 11 της συνθήκης. Η συνθήκη προβλέπει συνεργασία επί της ουσίας στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε πέντε χρόνια το πολύ από τη στιγμή που αρχίζει να ισχύει. Η ανακοίνωση παρουσιάζει επίσης διάφορες εναλλακτικέ για το συντονισμό αυτό. Όσον αφορά τώρα την ερώτησή σας για την φύση των συμβατικών διακανονισμών στα πλαίσια του μέσου ανταγωνιστικότητας, βασιζόμαστε στη συνθήκη και οι συμβατικοί διακανονισμοί βέβαια θα είναι πολιτικού χαρακτήρα. Οι σημερινές συνθήκε δεν προβλέπουν τη δυνατότητα νομικά δεσμευτικών τέτοιων ε, μέτρων. Θα πρέπει να υπάρχει απλώς συστήριξη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για την ερώτησή σας τώρα για το ποιες μεταρρυθμίσεις θα αποτελέσουν ε, προτεραιότητα, το μέσο αυτό θέλει να συνεισφέρει αποτελεσματικά για την καλή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και αυτό θα γίνει εφόσον τα κράτη-μέλη δεσμευθούν ακόμα περισσότερο να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις. Και εμείς θα στηρίξουμε τα κράτη-μέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα έχουν σαν αποτέλεσμα να υποφεληθούν και τα κράτη-μέλη μεμονωμένα αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιε μεταρρυθμίσει μπορεί να έχουν σημαντικέ επιπτώσει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και περιμένω τώρα τι απόψει σα για τι μελλοντικέ νομοθετικέ προτάσει όσον αφορά την ΟΝΕ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι ομιλητέ εκ μέρου των πολιτικών ομάδων πρώτα. Και ο πρώτο εκ μέρου του ΕΛΚ για τέσσερα λεπτά είναι ο κύριος Κοζές, ο αγαπητός συνάδελφος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ τίθενται κάποια ερωτήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι εξαιρετικά σημαντικά. Δώσατε κάποια στοιχεία απαντήσεων. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουμε άποψη όσον αφορά την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα αυτών των προτάσεων και την οικονομική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσφατη ιστορία μας δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει με ταχύτητα. Παρόλα αυτά, οι αδυναμίες της οικονομίας, οι αδυναμίες της Ευρωζώνης είχαν πολύ αρνητικές επιπτώσεις, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν μέσα και εργαλεία τα οποία να μπορούν να επιτρέψουν δράση στοχευμένη. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συστηματική δυνατότητα αντίδρασης πέραν της διακυβερνητικής δάσης. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι επίγον, αγαπητοί συνάδελφοι, να επανέλθουμε σε κοινοτικά μέσα και εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε με αποτελεσματικό τρόπο και να έχουμε και μια προληπτική δράση που θα μας επιτρέπει να αποφεύγουμε αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, συγγνώμη, να εκφράσω εδώ τον θαυμασμό μας όσον αφορά την αποτελεσματική σας δράση και την αποφασιστικότητά σας. Είναι πολύ σημαντικό να οδηγηθούμε προς μια πραγματικά νομισματική και οικονομική ένωση στην Ευρώπη. Οι δεσμεύσεις του 2012 στο σχέδιο της Επιτροπής μετά από πρότρινση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι ευπρόσδεκτες. Στην επόμενη συνάντηση κορυφής ελπίζουμε, ελπίζουμε πραγματικά συγκεκριμένα μέτρα να προταθούν και να καθοριστούν. Βεβαίως οι στόχοι αυτοί είναι αξιοσημείωτοι. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ε, οικονομικής ολοκλήρωσης, αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία σε εθνικό επίπεδο και αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να προχωρήσει η Ευρώπη σε περισσότερη ανταγωνιστικότητα, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξη. Το θέμα είναι πώς αυτές οι προθέσεις θα γίνουν πραγματικότητα και γι' αυτό και αναρωτιόμαστε σήμερα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δεν πρόκειται να κάνω συγκεκριμένες επιπλέον προστάσεις εδώ θεωρώ ότι η συνεισφορά του Κοινοβουλίου είναι χρήσιμη και σημαντική. Και θα αναφερθώ απλώ σε κάποια σημεία. Συντονισμό των μεταρρυθμίσεων των οικονομικών πολιτικών. Αυτό είναι απαραίτητο. Τα εθνικά μέτρα σε τομείς που είναι ευρωπαϊκοί τομείς πρέπει να αποφεύγονται. Και αυτό το βλέπουμε με την πληθώρα τραπεζικών προτάσεων και νόμων, κάτι με το οποίο θα ασχοληθεί η Επιτροπή, πιστεύω το Σεπτέμβριο, με την μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Υπάρχουν βεβαίως μέτρα εθνικά, τα οποία σήμερα έχουν ληφθεί και τα οποία δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά μέτρα εθνικά τα οποία έχουν επιπτώσεις σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης που προϋποθέτει συμβατικές διευθετήσεις και διακανονισμούς ενώ πολλές φορές ε, χάνουμε τον πραγματικό μας στόχο που είναι να ανακτηθεί η μακροοικονομική ισορροπία. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε ότι δεν θα πρέπει να εκταμιεύονται κονδύλια εάν δεν υπάρχει προηγουμένως υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για τις οποίες έχουν δεσμευθεί τα κράτη-μέλη. Ο δημοκρατικός έλεγχος θα πρέπει να είναι προϋπόθεση. Τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν σε εθνικό επίπεδο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επαγρυπνεί για τον δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ πραγματικά ότι βρισκόμαστε σε μια πρώτη φάση εναρμόνισης των θέσεων στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε και την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ και να δημιουργήσουμε πραγματικούς δείκτες για να μπορούμε να αξιολογήσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ευχαριστούμε κύριε Κωσές. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών το λόγο έχει η κυρία Φερέιρα για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις διευκρινήσεις που δώσατε. Λυπάμαι όμως δεν ήσασταν αρκετά λεπτομερείς διασχίζουμε μία περίοδο όπου ε, χρήζουν διευκρίνηση σε όλες οι δηλώσεις μας. Συντονισμός εξάντε μας είπατε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα, ε, τη σήμερον ημέρα αυτό συνιστά εξαιρετικά ευρεία ερμηνεία των ενίων διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα, στον Ευρωπαϊκό Διάλογο ουσιαστικά αυτό συνεπάγεται επιβολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρων περικοπών των μισθών λιτότητας ε, και ε, πολλές φορές, ε, αν όχι πάντα θα έλεγα, δεν εκπλήρωσαν τους προδιαγεγραμμένους στόχους. Χρειαζόμαστε συνεργασία, ε, οφείλουμε να επανεισάγουμε τον κοινοτικό μηχανισμό για να επιτύχουμε τη σύγκληση και την συνοχή και να μην ασχολούμαστε μόνο με την ανταγωνιστικότητα. Το μηχανισμός τώρα που προβλέπεται αυτή τη στιγμή για την στήριξη της σύγκλησης και της ανταγωνιστικότητας ε, έχει το δυναμικό να αναδειχθεί σε ένα θετικό βήμα στο μέτρο όμως ε, που θα υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη σε σχέση με τις επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητα είναι μια ευρύτατη έννοια που εντάσσεται ήδη στην στρατηγική 2020 και σίγουρα δεν περιορίζεται στην περικοπή ε, των μισθών και τις εξωτερικές έξωθεν επεμβάσεις στην αγορά εργασίας. Ε, ε, περιορίζεται το περιθώριο ελιγμών των κρατών μελών, όλο και περισσότερο, κυρίως των μελών που είναι στην Ευρωζώνη. Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενε κοινωνικές πρακτικές διαβούλευσης. Αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό, όπως επίσης και κάποιες διατάξεις κοινωνικού χαρακτήρα. Ελίζα. Ευχαριστούμε πολύ, Λίσα. Έχει περάσει ο χρόνο. Έτσι, έχει ξεπεραστεί ο χρόνο σου. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Γκουλάρ, εκ μέρου των φιλελεύθερων. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Όπω το είπε και ο Ζαμπόλ έτσι και εγώ θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει το έργο σα και η αποφασιστικότητά σα μεταξύ των επιτρόπων απέναντι στα κράτη-μέλη. Η απάντησή σα προσπαθεί να είναι βέβαια ισορροπημένη. Υπάρχουν ε, δύο σημεία πάρα πολύ θετικά. Το πρώτο είναι ότι λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση που έχει κάθε απόφαση κρατών μελών. Ο εξάνατος συντονισμό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μέχρι τώρα είχαμε ένα ενιαίο νόμισμα, αλλά με διαφορετικές ε, οικονομικές πολιτικές, κάτι το οποίο ήταν καταστροφικό για τους υπόλοιπους. Το δεύτερο θετικό είναι η δυνατότητα αυτή αλλά καρτ να αποφασίζουμε με τα διάφορα δημοσιονομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να προχωρήσουμε υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Συγχρόνως όμως υπάρχουν και δύο πράγματα που με απασχολούν και που εντοπίσαμε στο κείμενο και τα υπογραμμίζω τώρα. Πρώτον, θα δυσκολευτείτε γιατί εξ ορισμού ε, δεν αρέσει σε όλους η κοινοτική μέθοδος. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο οργανώνεται ανά χώρα. Προσοχή λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτό. Έχουμε δηλαδή λιγάκι την αίσθηση, κοιτώντα τα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια, ότι πολλά προτείνονται, πολλά ανακοινώνονται, αλλά οι πολίτες δεν τα νιώθουν στο πετσί τους πάρα πολύ αργότερα, όπως έγινε με την νομοθετική δέσμη των 2, 6 μέτρων κλπ. Προσοχή λοιπόν. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε νομοθετικό επίπεδο. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με πολίτες οι οποίοι δεν μπορεί να είναι όμοιροι της χώρας μέσα στην οποία γεννήθηκαν ή ζουν. Οπότε οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει διάκριση για, τους, ε, για τους πολίτες. Και βασιζόμαστε σε εσά για να φροντίσετε να λυθεί και αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε κυρία Γκούλαρ. Εκ μέρους των πράσινων τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γκίγκολτ. Δύο λεπτά, δυόμιση λεπτά παρακαλώ, κύριε Γκίγκολτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Είναι κρίμα γιατί δεν είναι παρόν το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είναι το επίκεντρο αυτής της συζήτησης. Κάτι που φυσικά δεν μας αρέσει πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει το δημοσιονομικό σύμφωνο είναι κάτι που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει ανοιχτά λίγο πολύ έχει εκφραστεί η δυσπιστία στο θέμα αυτό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρόταση καθότι πέραν των μέσων και των εργαλείων που προτείνονται είναι ξεκάθαρο πλέον το ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Κάτι που μου φαίνεται επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι επιγόντως χρειαζόμαστε περαιτέρω νομοθετικά μέτρα έτσι ώστε η βάση στην οποία βρίσκονται όλα αυτά τα εργαλεία και τα μέσα που διαθέτουμε να μας ε, κάνουν να συνειδητοποιήσουμε ότι ναι, έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα, δεν έχουμε όμως ε, τις απαραίτητες ε, διευκολύνσεις και διαδικασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιέσεις και τάσεις στην οικονομία, τον πληθωρισμό και άλλες απειλές οι οποίες σήμερα ε, χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι λοιπόν μια σοβαρή προσπάθεια να δώσουμε περισσότερη εργασία στους άνεργους της Ευρώπης, μια ενίσχυση του προϋπολογισμού, μια μακροοικονομική ισορροπία, όλα αυτά τα θέματα τα οποία βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των ανησυχιών μας. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τον κοινωνικό πυλώνα, κάτι το οποίο επίσης ε, είναι στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Τα διάφορα σχέδια τα οποία βλέπουμε σήμερα, σχέδια νομοθεσίας, θα πρέπει να υλοποιηθούν, θα πρέπει να γίνουν πράξη και τα δύο εργαλεία τα οποία συζητούμε σήμερα είναι ίσως τα πιο ζωντανά στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, θεωρώ ότι ο συντονισμός εξάντε κάτι που δεν υπάρχει πλέον από ό,τι καταλαβαίνω εγώ στον Συμβούλιο, πώς μπορούμε να τον επαναφέρουμε, να τον ενδυναμώσουμε επίσης όσον αφορά το CCI. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι πλέον ξεκάθαρη, σαφέστατη. Και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινοτικής μεθόδου η ατζέντα για το 2020 είναι σαφής. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτού του είδους οι διευθετήσεις, οι συμβατικές και οι διακανονισμοί να βρεθούν εκτός της κοινοτικής δράσης. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά ο κύριος Έπινγκ τώρα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Αυτό όμω θα μας οδηγήσει σε μια σχεδιασμένη οικονομία με τον εξάντε συντονισμό μεγάλων οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φτάνει να γίνει ένα γραφείο σχεδιασμού, οικονομικού σχεδιασμού. Δηλαδή υπό τις Βρυξέλλες θα αποφασίζονται όλα και ο κύριος Ρεν βέβαια μπορεί να είναι πολύ καλός σε σχέση με τους σοβιετικούς ηγέτες, αλλά στο ίδιο αποτέλεσμα θα καταλήξουμε με τις πολιτικές αυτές. Μια ε, οικονομική ένωση πρέπει να επιβιώνει. Εμείς προσπαθούμε να την διορθώσουμε. Υιοθετήσαμε τη δέσμη των δύο, τη δέσμη των έξι μέτρων. Εγώ τα υπερψήφισα. Τώρα όμως θέλουμε να σχεδιάσουμε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομική. Η οικονομία όμως εξελίσσεται βάσει ανταγωνισμού και οικονομικής ανάπτυξης, όχι βάσει σχεδιασμού. Ο κύριος Αντόρ πρόσφατα είπε ότι η Γερμανία πρέπει να αυξήσει τους μισθούς. Σύμφωνα με αυτόν, είναι υπερβολικά ανταγωνιστική η Γερμανία. Πρέπει να μειώσει την ανταγωνιστικότητά τη για να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο με του υπόλοιπου στην Ευρώπη. Άρα, δηλαδή, ο κεντρικό αυτό σχεδιασμό τι σημαίνει. Σημαίνει ισοπαίδωση όλων και όχι δυνάμεις της αγοράς. Πού θα οδηγηθούν τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία απλώς θα ενημερώνονται όχι, κύριε Ρέντε, συμφωνούμε. Νομίζουμε ότι θα έπρεπε να μπορούν να ψηφίζουν για του μηχανισμού. Ο κεντρικό αυτό οικονομικό σχεδιασμό δεν θα λύσει και τα προβλήματα του ευρώ. Αντίθετα, θα μα οδηγήσει σε πιο μεγάλη ύφεση ακόμα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι η Ευρωζώνη είναι μια αποτυχία έτσι όπω έχει σήμερα, ότι ήταν ιστορικό λάθο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτή την κατάσταση, να δει άλλου μηχανισμού οι οποίοι θα ε, μπορούν ε, να κάνουν εφικτό το να αποσυρθεί μια χώρα από την Ευρωζώνη. Να υπάρχει ελαστικότητα στο σύστημα αυτό, ευελιξία. Κάτι το οποίο βέβαια μισούν όσοι κάνουν κεντρικό σχεδιασμό. Δεν θέλουν να παραδέχονται τα σφάλματα και αφήνουν γενιές ολόκληρες να βλέπουν το μέλλον τους να εξατμίζεται. Κύριε Ρεν, η περιστρόικα, αν δεν εφαρμοστεί και εδώ, θα είναι πολύ αργά και ο δικός σας κεντρικός σχεδιασμός θα πλήξει το μέλλον πολλών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Βότμαν Κόλ θέλει να ρωτήσει κάτι. Δέχεστε την ερώτησή σας. Παρακαλώ. Ερώτηση από την κυρία Βότμαν Κόλ είπατε. Ναι, ναι, βεβαίως. Η κυρία Βότμαν Κόλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είναι ντροπή ο κύριος Έπινγκ να συγκρίνει με τον Πρέσνιεφ τον Επίτροπο Ρεν ενώ ο κύριος Έπινγκ στήριξε την δέσμη των 6 μέτρων. Και ξέρουμε ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό και ο Επίτροπος Ρεν. Δεν μπορεί λοιπόν όταν έχουμε τέτοιες ε, συστάσεις, αντί να στηρίζει τον Επίτροπο Ρεν ο κύριος Έπινγκ, να κάνει το αντίθετο. Ο κύριος Έπινγκ έχει στηρίξει και τις μικρές χώρες και τις μεγάλες χώρες και έχει κάνει τις σωστές θέσεις. Αυτό δεν είναι πιο σημαντικό. Για πείτε μου κύριε Επίγκ. Κύριε Βόρτμαν Κόλ. Θα απαντήσω κι εγώ στα Ολλανδικά. Προσπάθησα να κάνω χιούμορ. Η σύγκριση με τον Μπρέσνιεφ έχει να κάνει μόνο με τον κεντρικό σχεδιασμό. Με τίποτα άλλο. Και έχω την εντύπωση ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Προ τα εκεί πάμε, προς τον κεντρικό σχεδιασμό. Ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φιλελεύθερο σχέδιο. Και πού πάει τώρα. Τα εθνικά κοινοβούλια πια δεν έχουν τίποτα να πούνε. Υπάρχει δυσαρέσκεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε όλους τους πολίτες. Λοιπόν, οι πολίτες αντιτίθενται σε αυτό το κεντρικό σχεδιασμό, κυρία Βόρτμαν Κόλ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Πίνγκ. εκ μέρους... Α, μια στιγμή. Εκ μέρους της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο κύριος Μπλουμ. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Α, δεν είναι όμως. Εδώ, στο ημικύκλιο, δεν τον βλέπω. Η Ελευθερία και η Δημοκρατία όμως είναι παρούσες εδώ στο ημικύκλιο, έτσι ανεξάρτητα από την ομάδα που φέρει τον τίτλο αυτόν, λέει ο πρόεδρο. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Κλούτε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα από προσωπικής απόψης να πω ότι πραγματικά είμαι πεπισμένο ότι μία πιο ισχυρή οικονομική ολοκλήρωση είναι απαραίτητη στην Ευρώπη. Αυτό όμως μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν υπάρχει ενίσχυση πολιτική και δημοσιονομική. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η επεξεργασία της μέχρι τώρα κρίσης στην Ευρώπη από το Συμβούλιο είναι αντικείμενο κριτικής και δικαίως και αυτό οδήγησε τους Ευρωπαίους πολίτες να χάσουν την εμπιστοσύνη τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χάσουν την αξιοπιστία τους. Βλέπουμε ότι η ανεργία έχει αυξηθεί παντού στην Ευρώπη και εάν θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την οικονομική ολοκλήρωση θα πρέπει πραγματικά προηγουμένως να βρούμε τρόπο να ανακτηθεί η χαμένη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι χωρίς αυτά τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην οικονομική ολοκλήρωση. Αυτή θα αποτύχει. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά με στενοχωρεί ιδιαίτερα. Είμαι Γερμανός και η ιστορία μου με οδηγεί σε μια στενή και πραγματική δέσμευση σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα και στην επιτυχία του. Αλλά πραγματικά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης να γίνει εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών και της κοινωνικής στήριξης και συνοχής. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εξαλειφθεί η κοινωνική πτυχή αυτής της πολιτικής. Ο κύριος Τσίλτσα έχει το λόγο. Για 1,5 λεπτό. Η εμβάθυνση στην ΟΝΕ είναι κάτι που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει, λέει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα μεταρρυθμίσεων των χωρών μελών πριν αυτά πάνε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει το δικαίωμα, αλλά την έγκριση αυτή δεν μπορεί να την απαιτεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια μετά από τη δικιά της την έγκριση. Και κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένο από μια τέτοια πρόταση, γιατί έτσι μειώνονται οι αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων, άρα των εκπροσώπων των πολιτών. Ποιος μπορεί να δεχτεί κάτι τέτοιο είναι κάτι για το οποίο έχουν αγωνιστεί τόσες χώρες για χρόνια και χρόνια και τώρα να καταργήσουμε αυτό το δικαίωμα. Εμείς θέλουμε περισσότερη δημοκρατία. θέλουμε να ενισχυθεί η δημοκρατία, ενώ την μειώνει η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Η, Euro, η Ευρωζώνη έχει αποδειχτεί ότι δεν έχει λειτουργήσει. Η Ευρωζώνη λοιπόν πρέπει να διαλυθεί και να ενισχυθεί η εθνική κυριαρχία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν από μόνα τους να αποφασίσουν τι θέλουν βάσει αυτού που ζητάνε οι πολίτες τους. Άρα χρειαζόμαστε λιγότερη ε, κεντρική εξουσία. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν αυτό να το υπογραμμίσουμε και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Τελειώσαμε με τις πολιτικές ομάδες εδώ και τώρα περνάμε στους συναδέρφους που ατομικά παρεμβαίνουν στη συζήτηση. Με πρώτον τον κύριο Μπροκ για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να διαπιστώσω ότι θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση εάν δεν υπήρχε το ευρώ. Σήμερα οδηγούμαστε σε περισσότερη αλληλεγγύη χάρη στο ευρώ και ουσιαστικά αποφύγαμε μία κρίση όπως αυτή του 1929 χάρη στο ευρώ. Βεβαίως όλα δεν είναι ρόδινα και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Θεωρώ προσωπικά ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ληφθεί σοβαρές αποφάσεις, έχουν αποφασιστεί εργαλεία και μέτρα, τα οποία ουσιαστικά μπορούν να μας επιτρέψουν να έχουμε μια κοινή δράση και μια κοινή αντιμετώπιση. Βεβαίως, έχουμε κατά κάποιο τρόπο χάσει τον συντονισμό μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτές οι δύο προτάσεις της Επιτροπής είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η διακυβερνητική δράση δεν αρκεί και χρειάζεται μια νομοθετική πρόταση σαν αυτή που μας κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να οδηγηθούμε σε περισσότερη κοινοτική δράση, κοινή δράση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστή η πρόταση του Προέδρου Ολόντ, γιατί ουσιαστικά οδηγεί σε περισσότερη διακυβερνητική δράση, σε διεύρυνση της διακυβερνητικής δράσης και περιορίζει την Ευρώπη στην Ευρώπη της Ευρωζώνης, των 17. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνει 27 κράτη-μέλη. Δεν πρέπει λοιπόν να οικοδομήσουμε νέα σύνορα και νέα εμπόδια. Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν ε, βάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα αποτελέσουν κατευθυντήριες γραμμές, προϋποθέσεις για τις μελλοντικές μας αποφάσεις. Οι συμβατικές διευθετήσεις και διακανονισμοί σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε επιπλέον κοινοβουλευτικό και δημοκρατικό κενό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε επίσης να μην ουσιαστικά δημιουργήσουμε νέες δομές, νέες διαρθρώσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν περισσότερη γραφειοκρατία. Πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Θέλουμε να οδηγηθούμε προς ανάπτυξη. Όταν αναφερόμαστε στους νέους και στην ανεργία των νέων, πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αρκεί να αναφέρουμε τους αριθμούς των άνεργων νέων στην Ισπανία. Χρειαζόμαστε πραγματικές διαδικασίες κατάρτισης επαγγελματικής, οι οποίες θα επιτρέψουν σε αυτούς τους ανθρώπους να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας. Πρέπει να οδηγηθούμε σε θετική ανάπτυξη και αυτό προϋποθέτει τις δομές αυτές που σήμερα λείπουν στην Ευρώπη. Και αυτό χρειάζεται επενδύσεις ιδιωτικές επενδύσεις, δημόσιες προσπάθειες. Ξεπεράσατε το χρόνο σας. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπροκ. Κύριε Μπροκ. Κύριε Μπροκ. Υπάρχει κάποιος Γερμανός από την ομάδα σας, ο κύριος Ρούμπικ, που θέλει να σας ρωτήσει κάτι, κάτι σπάνιο. Σπάνια συμβαίνει αυτό. Δέχεστε, είναι τιμή, ναι. Εντάξει. Θέλετε να τιμήσετε λοιπόν τον συμπατριώτη σας και συνάδελφό σας με την ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος είναι από τη Γερμανία και εγώ είμαι Αυστριακός. Πολλές ερωτήσεις λοιπόν μπορώ να του θέσω. Μία από αυτές είναι η εξής. Πιστεύετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ίδια ε, μέσα ίδιους πόρους έτσι ώστε αυτή η προσπάθεια διάσωσης να γίνει πιο αποτελεσματική και να φτάσουμε σε μια σταθερότητα. Πολύ θα με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψη του Έλμαρ Μπρόκ για αυτό το θέμα. Θεωρώ Έχετε το λόγο κύριε Μπροκ. Θεωρώ πραγματικά ότι όσον αφορά το δημοσιονομικό πολιετές ε, πλαίσιο και τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους, οι δυνατότητες και τα εργαλεία που διαθέτουμε είναι βεβαίως σημαντικά, αλλά σαφώς και θα πρέπει εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες. Το θέμα του ευρώ Κύριε Ρούμπιχ, έχετε δίκιο να το τίθετε σε αυτό το πλαίσιο, αλλά ακόμα προϋποθέτει πολλές δυνατότητες που δεν έχουμε. Ο κύριος Γκαλτιέρη. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ και υπάρχει σύγκληση. Θα συνοψίψω ποια είναι η σύγκληση αυτή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει συναπόφαση και να δούμε τι θα γίνει με τις ε, χώρες μη ευρώ. Πρόκειται για ένα μέτρο ενθάρρυνση, αλλά πρέπει να αποσαφινιστούν κάπως τα πράγματα. Μιλάμε για επιπλέον πόρους και όχι για μακροοικονομική ερεσιμότητα. Έπειτα, ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μέσα στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ε, χρηματοδότηση από ορισμένες χώρες μέλη κάτι το οποίο θα ενισχύσει την Ευρωζώνη. Τώρα, αντί για συμβάσει υποχρεώσει. Εμεί θέλουμε έναν κώδικα σύγκληση που να αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο συν εθνικό για αποφάσει οι οποίε λαμβάνονται στα κράτη-μέλη με την πλήρη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Στη συνέχεια, οι κοινωνικέ ανισότητε θα πρέπει να έχουν την ίδια σημασία όπω η ανταγωνιστικότητα των τιμών. Εμεί πιστεύουμε ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι λογική θα ληφθεί υπόψη και ιδιαίτερα ε, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μία ε, νομοθετική πρόταση και οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σήμερα στο Συμβούλιο δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν τα νομοθετικά προνόμια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που δεν θα πρέπει να περιμένει πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό τώρα το λόγο έχει η κυρία Λούνατσεκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο πέρασε χωρίς ε, να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και αυτό οδήγησε σε περισσότερη φτώχεια, περισσότερη δυσκολία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχουν διάφορες συμφωνίες και διευθετήσεις που γίνονται διμερώς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Και βλέπουμε ότι σήμερα ζητάμε εξοικονομήσεις και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυξημένη ανταγωνιστικότητα. Βλέπετε όμως ότι οι πολίτες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν σκληρά μέτρα και αδικία, άδικη επιβολή αυτών των μέτρων. Θέλουμε λοιπόν περισσότερη αλληλεγγύη, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των κρατών μελών, έτσι ώστε πραγματικά να πιστούν πάλι οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι αυτή η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη που έχει σαν σκοπό να τους εξυπηρετήσει. Είναι μια Ευρώπη με αλληλεγγύη. Ευχαριστούμε κυρία Λούνατσεκ και συγχαρητήρια στους διερμηνείς, λέει ο πρόεδρο που κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά του χωρί να πατήσουν το κουμπί για να μου ζητήσουν να σα πω να μιλάτε πιο αργά. Η κυρία Βίκη Φόρτο, για δύο λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Θα καταψηφίσουμε την πρόταση. Ξέρετε, δεν είμαστε όλοι στην Ευρωζώνη και στη χώρα μου είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται και να προσχωρήσουμε. Εγώ πιστεύουμε στην εθνική κυριαρχία και εγώ προσωπικά, οπότε δεν νομίζω ότι είναι δική, σας δουλειά, δική μας δουλειά να πούμε στις χώρες Ευρωζώνης τι θα κάνουν. Όμως, σε ορισμένα ζητήματα επηρεάζονται και οι χώρες που δεν μετέχουν στην Ευρωζώνη και άρα χρειάζεται συζήτηση. Λοιπόν, καλείτε για σύγκληση για ένα μηχανισμό σύγκλησης και ανταγωνιστικότητας. Ωραία. Αλλά αυτό μπορεί να συνεπάγεται μεταφορά χρημάτων φορολογουμένων από τη μία χώρα στην άλλη και μπορεί να αποτελέσει αυτό ένα νέο κομμάτι του προϋπολογισμού. Για ποιο λόγο πρέπει να ε, γίνει αυτό. Δεν μας ρώτησαν εμάς καθόλου. Μας ανησυχούν όμως οι επιπτώσεις πρότασης ε, εκτός Ευρωζώνης. Βάσει τι διαδικασίες του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου προβλέπεται ομόφωνη συγκατάθεση των 27 Εθνικών Κοινοβουλίων για το προϋπολογισμό και τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές κάθε 7 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι είναι υπέρογκο ο προϋπολογισμός ε, και εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να διωγγωθεί έτσι περαιτέρω. Νομίζω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια κάθε 7 χρόνια θα ε, μπορέσουν να επέμβουν και να φρενάρουν αυτούς που ζητούν ακόμη μεγαλύτερες ή υψηλότερες δαπάνες. Ε, ε, ζητάτε μηχανισμό εκ τόσο ορίων του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να γίνει αυτό, ε, ούτω, ώστε οι συναρμόδιες αρχές ε, για τον προϋπολογισμό να μπορέσουν να αποφανθούν. Εγώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παρακάμψει τις εθνικές κυβερνήσεις σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες ε, μέσω αυτού του μηχανισμού και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι χώρες της Ευρωζώνης κυρίως θεωρούν ότι έχουν απολέσει κάθε έλεγχο έχω κάθε εθνική κυριαρχία. Το Εθνικό Κοινοβούλιο πάντως δεν θα πρέπει να διωγγωθεί. Ένα λεπτό κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Πώς ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση μέσω μιας ιδεολογικής προσέγγισης. Αντί να αλλάξουμε την ιδεολογία και την πολιτική, κάνουμε το ίδιο ξανά και ξανά. Και περιμένουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Μα εξορισμού δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε κανένα αποτέλεσμα. Η υποχρέωση των κρατών μελών είναι να ακολουθήσουν την ίδια ιδεολογική προσέγγιση. Μα αυτή είναι μια συνταγή για σίγουρη καταστροφή στο μέλλον. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα επενδύσεων για να δημιουργούν νέε θέσει απασχόληση, για να ενισχυθεί το ΕΠΑ. Πού όμως είναι όλα αυτά, πώς αντιμετωπίζει η αποτυχία των τραπεζών, τι γίνεται με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που μας υποσχέθηκε ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πού είναι η έσχατη λύση δανεισμού. Μα η προσέγγιση που έχουμε μέχρι τώρα είναι η χειρότερη. Οι αποφάσεις οικονομικές παίρνονται από τα κράτη-μέλη χωρίς να υπάρχει μεταφορά πλούτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα όλα αυτά είναι οικονομικός αναλφαβητισμός στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Άντερσον. Δυόμιση λεπτά τώρα ο συνάδελφος Φέιο. Παρακαλώ κύριε Φέιο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε Επίτροπε, θα ήθελα αρχικά να σας ε, συγχαρώ για το μακρύ δρόμο που διασχίσατε από κοινού με το Κοινοβούλιο ε, για να θεσπίσετε την ε, Ευρωπαϊκή και Οικονομική Ένωση. Είδαμε το μηχανισμό ε, ανάπτυξης, είδαμε το μηχανισμό για τη ρύθμιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους δημοσιονομικού χαρακτήρα μηχανισμούς. Όμως, όλο ένα και περισσότερο και εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτό που μας ζητείτε είναι δημοσιονομική πειθαρχία ταυτόχρονα με την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά κατεπηγόντως αυτό μας ζητούν ε, οι πολίτες μας ε, και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή λύση και θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωσή της. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες ε, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η αναγκαιότητα συντονισμού των πολιτικών μας στον τομέα της οικονομίας και τη θέσπιση ενός μηχανισμού για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα θα ήθελα να γνωρίζω, Επίτροπε, αν με αυτά τα μέτρα θα μπορούσαμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εσωτερικό της Ευρωζώνης θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε επιτέλους ε, τις κυρώσεις ε, με τα απαιτούμενα κίνητρα προς τα κράτη-μέλη για να συμμορφωθούν. Εγώ είμαι από την Πορτογαλία και συμμορφωθήκαμε με αυτά που μας ζήτησαν. Όμως, ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και η επιβράβευση για τη συμμόρφωση στις συνέχεια με, ώστε οι πολίτες να συνειδητοποιούν ότι οι θυσίες που κάνουν αξίζουν τον κόπο. Αυτά τα κίνητρα και επιβράβευση δεν πρέπει να είναι κατά περίπτωση. Πρέπει με συστηματικό τρόπο να ενσωματώνονται στην κείμενη νομοθεσία. Ευελπιστώ ότι αυτό θα συμβεί και αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να περάσω σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι. Για 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Χουαγνό έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι ή που θα βγει από την παγίδα της λιτότητας και θα κάνει ένα άλμα προς τη δημοκρατία ή αλλιώς οι λαοί θα τη μισήσουν. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου έχει δώσει το χάρτη πορεία. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει τη δικιά τη δουλειά, ο Φρανσουά Ολόντ είπε ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή, αλλά δυστυχώ δεν ζητήθηκε η γνώμη του για την Κύπρο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έχει την Τρόικα απέναντι που αποφασίζει. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια κυβέρνηση χωρί κοινοβούλιο δεν σημαίνει δικτατορία. Το Κοινοβούλιο το υπενθύμησε επίση στην έκθεση Τάισεν ότι πρέπει να είναι παρόν σε όλα τα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στη συζήτηση που θα γίνει στου ελέγχου για τι ειδικέ ε, προτάσει αναχώρα. Πρέπει να είναι στην καρδιά του σχεδιασμού του ε, προπολογισμού στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό και μιλάμε για διμερείς σχέσεις ανάμεσα Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών που είναι κάτι το οποίο πρέπει να απορριφθεί. Δεν μπορεί να εφαρμόσουμε στην Ευρώπη μια τρόικα η οποία έχει αποδειχτεί λάθος σε όλη τη την πορεία. Είναι κάτι που πρέπει να καταργηθεί. Για να ενισχυθεί η διακυβέρνηση λοιπόν στην Ευρωζώνη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δικιά του δομή για την Ευρωζώνη, για τις χώρες εκείνες οι οποίε προσπαθούν να επιβάλλουν τα δικά του συμφέροντα απέναντι στα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, η δημοκρατία πρέπει να είναι στην καρδιά τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη των πολιτών και όχι μια Ευρώπη των συμβάσεων και των υποχρεώσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε. Ένα λεπτό τώρα ο κύριε, κύριε Φερέιρα. Ο κύριος Φεραίρα. ευχαριστώ πρόεδρε, επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση ήταν και παραεξακολουθεί να είναι το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου. Ε, μετά από δεκαετίες ε, του ευρώ βλέπουμε 36% ελλείψεις στους προϋπολογισμούς ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περικοπές στους μισθούς, επέμβαση στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε βεβαίως και θετικά αποτελέσματα του ευρώ, ταυτόχρονα όμως επιδεινώνεται η ποιότητα της ζωής, το βάρος των μισθών στο εθνικό εισόδημα μειώνεται, καταστρέφονται παραγωγικοί μηχανισμοί, από βιομηχανοϊοποιούνται χώρες ε, ε, και μετατρέπονται σε ε, χώρες καταναλωτές της παραγωγής των χωρών της κεντρικής Ευρώπης. Για ποιον ήταν όλα αυτά επωφελή. Θέλουμε να προχωρήσουμε και σε κάθε βήμα προς την ενοποίηση ότι προσπαθούν όλοι να νόμιμοποιήσουν τις παρελθούσες κινήσεις και τα μελλοντικά του σχέδια. Περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστούμε. Παύλο Σάλβαδη, δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όταν οικοδομήσαμε την Ευρωζώνη, ξέραμε ότι υπήρχαν κάποιες ατέλειες που οφείλονταν στο γεγονός ότι είχαμε μια ενιαία νομισματική πολιτική, αλλά όχι μια δημοσιονομική και οικονομική κοινή πολιτική. Κάτι το οποίο μας οδήγησε σε έλλειψη συντονισμού, η οποία ε, καταδείχτηκε ήδη από το 2005 στην έκθεση ΚΟΚ. Η κρίση του 2008 βέβαια ενίσχυσε τις ατέλειες αυτές. Ας είμαστε όμως θετικοί. Μας δόθηκε έτσι και η δυνατότητα όχι μόνο να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκολίες, αλλά και να βελτιώσουμε ολόκληρη την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Ευρωζώνη βγαίνουμε από την κλασική φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, προχωράμε βήμα-βήμα, στάδιο-στάδιο. Συμφωνούμε κάτι και το εφαρμόζουμε. Τώρα, επιστρέφουμε στην παλιά φιλοσοφία. Ένας από τους κύριους στόχους ήταν να δημιουργηθεί μια πραγματική οικονομική ένωση. Η Τραπεζική Ένωση αποτελεί μία πτυχή κατά προτεραιότητα που πρέπει να προωθήσουμε μέσα στην Οικονομική Ένωση. Όπως το λέγαμε και χτες εδώ στο Μικύκλιο. Ένα βήμα αποτελεί μόνο που δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει αλληλεγγύη. Μια αλληλεγγύη που δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτοματισμός αλλά που είναι αναγκαία βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Θέλω να συμφωνήσω με τον συνάδελφο και να υπογραμμίσω και εγώ την κοινωνική διάσταση που είναι αναγκαία. Αναγκαία και απαραίτητη. Χρειάζεται και ευελιξία, όπως πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης όπως σήμερα. Ο συντονισμός εξάντια των οικονομικών πολιτικών και το μέσο για το μηχανισμό σύγκλησης και ανταγωνιστικότητας είναι κάτι αναγκαίο για τις χώρες οι οποίες έχουν το ίδιο νόμισμα μεταξύ τους, αλλά που μερικές φορές, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν κοινό ορίζοντα, ενώ θα έπρεπε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ο εξάντες συντονισμός να εφαρμόζεται στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης και ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του για να προχωράει με μεταρρυθμίσεις. Συνεπώς ο μηχανισμός σύγκλησης και ανταγωνιστικότητας πρέπει να συνδυαστεί με έναν οικονομικό μηχανισμό, με στόχους, με προϋπολογισμό για να αντιμετωπιστούν τα σφάλματα του παρελθόντος. Τα δύο αυτά μέσα αποτελούν ένα βήμα παραπάνω τόσο αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή και Οικονομική Ένωση και εν τέλει και την Πολιτική Ένωση. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η απόφαση αυτή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Παύλο. 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το ξεπέρασμα αυτής της ε, ύφεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μέτρα που θα μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Δυστυχώς, εδώ βλέπουμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια περισσότερης ευελιξίας ε, στην αγορά εργασίας και αυτό είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Θα έπρεπε να μειωθούν οι διαφορές το έγγραφο της Επιτροπής ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποιες μεταρρυθμίσεις για περισσότερη λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις, ε, αποδυνάμωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και περισσότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε ότι η διαδικασία που επικράτησε στις Ηνωμένε Πολιτείες στηρίζει τέτοιες προσπάθειες στην Ευρώπη. Δεν είναι όμως αργά για να επανέλθουμε στην σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να τεθεί ο κοινωνικός πυλώνας στο επίκεντρο όλων των οικονομικών πολιτικών στην Ευρώπη. Περισσότερη αλληλική με κοινέ εγγυήσει για τα δημόσια ελλείμματα. Αυτό είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ, Τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Σάντσες Πρεθέσο. Πρόεδρε, πώς συμπεριφέρεται η ευρωπαϊκή οικονομία. Τα κράτη-μέλη προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις για το Σύμφωνο σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πετύχει του στόχου της Λισαβόνα και η Ευρώπη τελικά ανταποκρίνεται χειρότερα από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο στις προκλήσεις της κρίσης. Οι διακρίσεις έχουν οδηγήσει σε απώλειες θέσεων σε οικονομικές δυσκολίες του κόσμου, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΟΝΕ θα πρέπει να αναλάβει ευθύνη και να δείξει αλληλεγγύη, πειθαρχία αλλά και κίνητρα. Να πάμε στον οικονομικό συντονισμό εξάντε είναι κάτι θετικό, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο κοινή οικονομικής πολιτικής. Επίσης χρειάζεται και μια πολιτική κινήτρων για επενδύσεις. Στα πλαίσια αυτά της κοινή οικονομικής πολιτικής να ευθυγραμμιζόμαστε και με τους στόχους του 2020 υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Αλλά για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα ε, πολύ πλευρή, χρειάζεται συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να βασίζεται σε ένα κοινωνικό σύμφωνο και να πάμε πιο πέρα από τα μέτρα προβλέπονται στις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές με δημοκρατικό έλεγχο για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζονται πρωτοβουλίες στον τομέα ε, των πιστώσεων για να βελτιωθούν τα δημοσιονομικά των χωρών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Τέλειωσε ο χρόνος σας. Τώρα, το λόγο έχει ο κύριος Μπλουμ, ο οποίος έπρεπε να είχε πάρει το λόγο εκ μέρους της πολιτικής του ομάδας νωρίτερα. Αλλά δεν ήταν τότε, όταν ήταν η σειρά του, θα πάρει τώρα το λόγο. 1,5 λεπτό. Παρακαλώ κύριε Μπλουμ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ε, ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν ε, εδώ στην ώρα μου. Ξέρετε ότι δεν το συνηθίζω και σας ευχαριστώ ε, για την ευγενή καλοσύνη μου. Δίνετε το λόγο Κοίταξτε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα από τα βασικότερα ζητήματα όταν συζητείτε το ευρώ είναι η συνωμοσία και το κουκούλωμα. Αυτές είναι οι δύο λέξεις ε, κλειδιά πρόκειται γι' αυτό. Και ξέρετε, στην ε, Αγγλία δεν είμαστε σίγουροι τι συμβαίνει. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν μία αμυδρά, έστω και αμυδρά ιδέα περί οικονομικών, θα συνειδητοποιούν ότι αυτό το κοινό νόμισμα ήταν καταδικασμένο σε αποτυχία εξ αρχή ε, στο βαθμό που δεν συνοδευόταν από μία δημοσιονομική πολιτική. Χρειάζεται αυτή για να έχουμε ενιαία ισοτιμία και ενιαίο νόμισμα. Είναι μέρο του ίδιου πακέτου και ε, πώ να σα πω, εντάσσεται στο ίδιο οικονομικό φαινόμενο. Οι ε, θεωρίε λένε «Α, ήξεραν ότι θα συμβεί αυτό, το ήξεραν ότι θα καταρρεύσει το σύστημα το ήξεραν ότι αυτό θα συνεπαχθεί προβλήματα και βάσανα για χώρες που είναι αρκετά ανόητες ε, ώστε να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο μηχανισμό. Τι συμβαίνει όταν ε, καταραίει, όταν παίρνουν όλα φωτιά, όταν όλα πάνε κατά διαόλου, ε, τότε θα έπρεπε να πούνε ότι εκείνοι είναι οι συνομότες οι οποίοι προώθησαν ένα μη δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνηση και τον επέβαλαν στους ανθρώπους παρά τη θέλησή τους. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Αυτό είναι και η ουσία του σημερινού κειμένου. Αυτό περί αυτού πρόκειται. Είναι η απαρχή μια μη δημοκρατική διαδικασία, ούτω ώστε οι εκλογεί να αποκλειστούν από το σύστημα και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ευχαριστούμε. Τώρα ερχόμαστε στο Catch the του Πρόεδρου. Α, υπάρχει ερώτηση. Κύριε Μπλουμ, δέχεστε την ερώτηση της συναδέρφου μας. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο για την ερώτησή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε στην αρχή της παρέμβασής σας, κύριε Βλουμ, ότι απέτυχε η ΟΝΕ εφόσον δεν υπάρχει δημοσιονομική πολιτική και κίνητρα για συνεργασία. Πράγματι, γι' αυτό πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που, εκφράζουμε που δημιουργούμε τώρα συστήματα για να συντονιστεί η οικονομική μας πολιτική. Θέλουμε πιο κοινή προσέγγιση. Λοιπόν, δεν συμφωνείτε ότι τώρα βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Όσον αφορά την έλλειψη δημοκρατίας, Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να τα βάζουμε σε αντιπαράθεση. Χρειάζονται και τα δύο για τη δημοκρατία. Κύριε Μπλουμ, απαντήστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει κανεί, έτσι δεν είναι. Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική δημοσιονομική πολιτική, διότι δεν τέθηκε στους λαούς με δημοψήφισμα, ούτε με κανένα άλλο τρόπο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, μα το υποσχέθηκαν το δημοψήφισμα, αλλά στην πραγματικότητα εδώ και χρόνια μα το αρνούνται. Οπότε εγώ για το Ηνωμένο Βασίλειο μιλάω και λέω ότι δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτό. Δεν μπορεί λοιπόν να πιέσει κανεί για κοινή δημοσιονομική πολιτική. Για ρωτήστε τον κόσμο, είτε πρόκειται για την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, ρωτήστε του και θα πάρετε την απάντηση. Ευχαριστούμε κύριε Μπλουμ. Κάτσε λοιπόν. Η κυρία Παπαδοπούλου, ένα λεπτό παρακαλώ. Αντιγόνη, έχει το λόγο. Έχω την αίσθηση πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurogroup και η Ευρωζώνη είναι δυστυχώ ουραγή των εξελίξεων. Στο επίκεντρο των εξελίξεων είναι δυστυχώ η Τρόικα, η οποία δεν είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένη, δεν λογοδοτεί ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε σε Εθνικό Κοινοβούλιο, επιβάλλει αυστηρέ πολιτικέ λιτότητα στι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου, χωρί ανάπτυξη, χωρίς επενδύσεις και ουσιαστικά καταστρέφει τους λαούς οικονομικά και κοινωνικά και δείτε ένα απλό παράδειγμα η περίπτωση της ελλάδας και της κύπρου. για την περίπτωση της κύπρου κύριε olli θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ήρθε να κάνει εκ των υστέρων μια νεκροψία διότι ήταν λανθασμένες οι πολιτικές του eurogroup και δυστυχώς άδικη και πρωτοφανής η απόφαση για κούρεμα καταθέσεων. και διερωτούμε μόνο με νομοθετήματα θα μπορούσαμε να, διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και το eurogroup. εγώ θέλω μια απάντηση πώ στηρίζονται σήμερα οι πολίτε τη κύπρου και αυτό δεν μπορεί να γίνει με μελλοντικά νομοθετήματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σα στην συζήτηση αυτή, την τόσο ουσιαστική. Θα αρχίσω με το εξή. Συμφωνώ με τον κύριο Κοζές, τον κύριο Φεραίρε, τον κύριο Κιγόλτ και τον κύριο Κλούτε που υπογράμμισαν τη σημασία που έχει η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της οικονομίας, της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και της ΟΝΕ. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταση εξάλλου σε λίγα λεπτά. Δεύτερον, όσον αφορά αυτά που είπαν η κυρία Γκουλάρ και ο κύριος Μπροκ για την κοινωτική μέθοδο, η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στην κοινοτική μέθοδο επειδή πιστεύουμε από την εμπειρία μας ότι είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε μια πραγματικά βιώσιμη πολιτική και πραγματική πρόοδο δημοκρατικά, ώστε να υπάρχει πολιτική λογοδοσία. Αυτό σημαίνει ότι τα διακυβερνητικά μέσα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κοινοτικό πλαίσιο. Υπογραμμίζω επίσης μετά από αυτά που είπε η κυρία Φόρτ ότι με τις εξελίξεις της ΟΝΕ πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει η αικαιρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη. Υπογραμμίζουμε επίσης ότι για μας η βασική αρχή όσον αφορά το μέλλον της ΟΝΕ είναι ότι οποιοδήποτε βήμα υπερενισχυμένης αλληλεγγύη και αμοιβαιότητα των χρεών είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνοδεύεται με αυξημένη υπευθυνότητα. Δηλαδή να μοιραζόμαστε περισσότερο την κυριαρχία και την ακαιρεότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Κουλάρ αναφέρθηκε και στον κατακαιρματισμό των συστάσεων. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι κάνουμε τη σύσταση και στην Ευρωζώνη για τους λόγους που είναι προφανείς. διότι υπάρχει αλληλοεξάρτηση μεταξύ των χωρών μελών και ό,τι συμβαίνει στη μία χώρα επηρεάζει αυτά που συμβαίνουν στην άλλη. Το Eurogroup λοιπόν πρέπει να μπορεί να συζητήσει ποιο είναι το καλύτερο μείγμα πολιτικής προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία μας και να έχουμε ε, ανάπτυξη για το μέλλον. Κύριε Κιγκόλ, όσον αφορά τις συζητήσεις στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο περιμένω να συζητήσει τώρα τον εξάντε συντονισμό των μεγάλων οικονομικών μεταρρυθμίσεων και το θέμα των μηχανισμών αλληλεγγύης. Στη συνέχεια θα πρέπει, ελπίζω, να μας δώσει μια επικοδομητική και θετική απάντηση. Τέλος, Πρόεδρε, ένα σχόλιο προς τον κύριο Έπινγκ. Συχνά κάνει χιούμορ με τους λεκτικούς του ακροβατισμούς. Αυτή τη φορά με σύγκρινε με τον Μπρέσνιεφ. Η σύγκριση αυτή είναι λανθασμένη και ακατάλληλη πιστεύω. Είναι κακού γούστου το χιούμορ αυτό. Δεν έχετε καμιά άλλη ιδέα, δεν έχετε τίποτα καλύτερο να πείτε από αυτό. Έχω αρκετούς συγγενείς που έχουν χάσει τη ζωή τους γιατί πλήρωσαν με τη ζωή τους το τίμημα της ελευθερίας. Είμαι λοιπόν κατά του ολοκληρωτισμού και υπέρ της δημοκρατίας. Ο παππούς μου πέντε χρόνια ήταν στο μέτωπο και μου είπε μετά την εμπειρία του αυτή το χειμώνα εκείνο στον πόλεμο ότι πέρασε πέντε χρόνια κοιτώντας προς την Ανατολή ενώ έπρεπε να κοιτάω προς την Δύση. Εγώ κοιτάω και προς Ανατολές και προς Δυσμάς. Και γι' αυτό και συμφωνώ με τον κύριο Κλούτε με τα σοφά του λόγια, πιο σοφά από τα δικά σας κύριε Έπιγκ, που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί ως ένα σώμα υπέρ της ειρήνης και της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό όσον αφορά τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ. Έχω να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις από τους εισελιστές μου.